Good morning, everybody. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχίζουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση, η οποία θα κρατήσει μέχρι τις 12 και 4 σήμερα. Υπάρχει μια μικρή αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Το σημείο 5, η ψηφοφορία δηλαδή για το σχέδιο έκθεσης όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου έχει αναβληθεί για την επόμενη συνεδρίαση. Συνεπώς η έκθεση αυτή Χολμάιερ κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφιστεί στις 27 του μηνός και όχι σήμερα. Αν συμφωνείτε λοιπόν και δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για την τροποποίηση αυτή, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Επίσης, δυστυχώς σήμερα δεν έχουμε διερμηνία στα κροατικά, τα τσεχικά, τα μαλτέζικα, τα λετονικά, τα λιθουανικά, τα δανέζικα, τα εστονικά, τα σλοβενικά και τα γκέλικ. Έγκριση των πρακτικών. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις επί των ε, πρακτικών της 22ης 23ης Σεπτεμβρίου 2015 και της 20ης 6 Μαΐου 2016 θεωρούνται εγκεκριμένα. Εγκρίνονται συνεπώς και ερχόμαστε τώρα στο πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, το πρώτο ουσίας, που είναι η δεύτερη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την υλοποίηση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Στις 20 Απριλίου του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη της έκθεση όσον αφορά την υλοποίηση της ε, συμφωνίας και μας, ε, μας παρουσίασε την έκθεση αυτή εδώ στην ΛΥΜΠΕ, η Επιτροπή. Στις 9 Μαΐου είχαμε μια προφορική δήλωση της νομικής υπηρεσίας όσον αφορά την φύση της συμφωνίας. Και σήμερα καλωσορίζουμε εδώ τον κύριο Μορντου που είναι διευθυντή για την πολιτική και στρατηγική διεύρυνση όσον αφορά την Τουρκία τη DG NIR τη Επιτροπή, για να μα παρουσιάσει τη δεύτερη έκθεση προόδου για την υλοποίηση τη συμφωνία αυτή. Οπότε θα ακούσουμε πρώτα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους για συζήτηση. Παρακαλώ κύριε Μορντού, έχετε το λόγο. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα. Όπως λέει και ο τίτλος μου, εγώ ασχολούμαι κυρίως με τις δηλώσεις όσον αφορά την υλοποίηση τη συμφωνίας μας με την Τουρκία. Ήμουνα παρόν από την αρχή της χρονιάς, έχω πάει 20 φορές, προσπαθώντας να δω ότι η συμφωνία αυτή πράγματι υλοποιείται και προχωράει καλά προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο όντως έχουν προστασία όλα τα άτομα τα οποία χρήζουν προστασίας ε, εκεί. Θα σας πω δύο λόγια και μετά καλύτερα να αφήσουμε περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση. Θα αρχίσω λοιπόν λέγοντάς σας τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Η έκθεσή μας λέει ότι η κατάσταση βελτιώνεται αλλά είναι εύθραυστη ακόμα. Για να το δούμε από πλευρά της Τουρκία όσον αφορά το τι έχει κάνει η Τουρκία μέχρι τώρα. Στην έκθεσή μας λέμε ότι η Τουρκία πράγματι έχει αναλάβει σημαντικά βήματα τόσο νομοθετικά όσο και άλλα. Για παράδειγμα την εξασφάλιση των Συρίων αλλά επίσης και των μη ε, Συρίων μετά τις 4 Απριλίου όταν αυτοί επιστρέφουν που μπορούν να καταγραφούν για προσωρινή προστασία και να ζητήσουν διεθνή προστασία. Οι Τούρκοι επίσης έχουν επεκτείνει και το άνοιγμα της αγοράς τους εργασίας που περιοριζόταν στους Σύριους μόνο. Τώρα υπάρχουν αντίστοιχες διατάξεις και για άλλους και για η ίδια προστασία δηλαδή προσωρινή που δίνεται για τους Σύριους δίνεται και για τους μη Σύριους. Βλέπουμε επίσης και τις πρώτες επιπτώσεις μετά την χρηματοδόση, τη χρηματοδότηση που δώσαμε στην Τουρκία. Όπως ξέρετε, 3 δισεκατομμύρια περίπου δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα 740 εκατομμύρια ε, δίνουμε. 140 ήδη έχουν ε, δοθεί και δουλεύουμε με ένα χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε μέχρι το καλοκαίρι δύο δισεκατομμύρια να έχουν ε, δοθεί με πρώτα ένα και μερικά από τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η Τουρκία καλύπτονται από τα ποσά αυτά. Επιτόπου θέλουμε να δούμε τη διαφορά. Για παράδειγμα όσον αφορά τα παιδιά που πάνε σχολείο, που μπορούν να αποφεληθούν δηλαδή από τις σχολικές ε, ε, διευκολύνσεις, γιατί υπάρχουν κάπου 305.000 που δεν πάνε. Αν δούμε λοιπόν τα ποσά και ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση, τα τελευταία που ξέρω από χτες δηλαδή, μας παρουσιάζουν αρκετά καλά την κατάσταση από χτες το βράδυ. 8.390 πρόσφυγες είναι στα νησιά. Τι σημαίνει αυτό για τα συνολικά ποσά. Σημαίνει ότι από τότε που άρχισε η συμφωνία, κατά μέσο όρο κάθε μέρα κάπου 104 ε, περνάνε καθημερινά. Μέσα σε ένα μήνα, τον ολόκληρο προηγούμενο, το βλέπετε ότι τον Μάιο είχαμε 40 την ημέρα κατά μέσο όρο. Ενώ προηγουμένως πριν αρχίσει η ενεργοποίηση της συμφωνίας αυτής, από την 1η Φεβρουαρίου για παράδειγμα μέχρι τις 20 Μαρτίου, ο μέσος όρος στην περίοδο αυτή ήταν πάνω από 1630 πρόσφυγες που πέρναγαν ε, προς τα νησιά την ημέρα. Αν δούμε και πόσοι μετανάστες τώρα έχουν επιστρέψει στην Τουρκία, και αυτό είναι ενδιαφέρον, βλέπουμε συνολικά από χτες το βράδυ 468 μετανάστες έχουν επιστραφεί μέχρι χτες το βράδυ. Έτσι. Και αυτό σημαίνει ότι ήταν 31 Σύριοι, λίγοι δηλαδή σχετικά είναι οι Σύριοι. Όσον αφορά τώρα το θέμα της μετεγκατάστασης, εδώ βλέπουμε από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 711 και 370 ακόμα περιμένουν για να μεταγκατασταθούν από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω όμως εδώ να υπογραμμίσω κυρίως ένα πράγμα και εδώ γίνεται πολλή συζήτηση για τα θετικά και τα αρνητικά της συμφωνίας. Ένα πάντως που θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι αν δούμε για τους θανάτους, τι θανάτους είχαμε τον Ιανουάριο μόνο, κάπου 70 μόνο τον Ιανουάριο, από τότε που ισχύει η συμφωνία έχουμε 7 συνολικά και κανέναν το Μάιο θάνατο. Παρά τις επικρίσεις λοιπόν, αξίζει να πάρει κανείς κάποια απόσταση και να διαπιστώσει ότι έχει κάνει τη διαφορά, ότι έχει μειωθεί αυτή η απώλεια ανθρώπινων ζώων που είχαμε πριν. Κατά τη γνώμη μου επίσης, αρκετά αποτελεσματικά διαλύονται και τα δίκτυα των ε, ανθρώπων που υποφελούνται και λαθρέα περνούσαν τους πρόσφυγες, οι λαθροδιακινητές. Τα δίκτυά τους έχουν καταστραφεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Δεν είναι όπως πριν από ένα χρόνο. Η αγορά αυτή, εντό εισαγωγικών όσον αφορά το Αιγαίο, έχει διαλυθεί. Μπορούμε να εκφράσουμε πλήρη ικανοποίηση. Όχι, δεν νομίζω. Κυρίως αν κοιτάξουμε τις επιστροφές που έχουμε προς την Τουρκία από τότε που άρχισε να υλοποιείται η συμφωνία. Εξακολουθούν να είναι χαμηλά τα νούμερα. Είπα πριν 766 έχουν επιστραφεί που σημαίνει ότι τα hot spots στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι πολύ φορτωμένα. Ο κύριος λόγος που το νούμερο αυτό δεν είναι υψηλότερο έχει να κάνει με όλους εκείνους τους παράτυπους μετανάστες που φτάνουν στην Ελλάδα και που είναι από άλλες εθνικότητες όπου δεν αναγνωρίζεται γενικά το δικαίωμά τους στο άσυλο. Παρόλα αυτά έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου. Και πρέπει να ξέρετε ότι κάθε αίτηση ασύλου εξετάζεται σε ατομική βάση. Το έχω ξαναπεί εδώ. Όντω αυτό γίνεται. Και πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η συμφωνία υλοποιείται σεβόμενη πλήρως το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο που δίνει τη δυνατότητα να υποβάλει κανείς αίτηση για άσυλο. Γι' αυτό λοιπόν οι επιστροφές δεν είναι πάρα πολλέ. Ο μεγαλύτερος αριθμός ε, αιτήσεων λοιπόν που έγινε κατέληξε στο γεγονός ότι έχουν δικαίωμα σε άσυλο. Αυτές που δεν ε, κρίνονται ως αποδεκτές έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν, να κάνουν κάποιο είδους έφεση. Και οι ελληνικές αρχές μετά από την πρώτη απάντηση εξετάζουν εκ νέου τις αιτήσει αυτές. Κάτι που σημαίνει ότι οδηγούμαστε σε καθυστερήσεις, γιατί πρέπει να κάνουν δύο φορές τη δουλειά. Και οι περισσότερες αποφάσεις μέχρι τώρα και τα οι αρχές οι οποίες ασχολούνται με τη δεύτερη εξέταση καταλήγουν πάλι πολύ συχνά στο ότι δεν είναι παραδεκτές οι αιτήσει αυτές. Πάντα όμως επιμένω ότι το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο προβλέπει κατά περίπτωση εξέταση της αίτηση ασύλου. Οπότε κάθε φορά που γίνεται κάποιο είδους έφεση πρέπει να γίνει πάλι ατομικά. Μας πήρε χρόνο, όπως είπα και πριν, προκειμένου στην Ελλάδα να έχουμε όλες τις διαδικασίες ώστε να συνοδεύονται οι διατυπώσεις αυτές. Τώρα περιμένουμε πιο γρήγορα να προχωρήσει η επεξεργασία των αιτήσεων και έτσι πολύ πιο γρήγορα όλοι αυτοί οι παράτυποι μετανάστες να επιστρέψουν στην Τουρκία. Όσον αφορά τώρα τους χώρους όπου γίνεται η επεξεργασία αυτή, η Λέσβος, η Χίος και η Σάμος έχουν αποφορτιστεί κάπως τα hot spots εκεί. Στην ε, επίση υπάρχουν ε, χώροι που εκπαιδεύουμε τον κόσμο για να μπορέσει να επεξεργάζεται όσο γίνεται πιο γρήγορα και όσο γίνεται περισσότερες συνεπώς αιτήσει για άσυλο. Οι ελληνικές αρχές εκ παραλίλου σε συνεργασία με την IOM και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει ένα πρόγραμμα εθελοντικών επιστροφών. Και αν δείτε πόσοι τελικά έχουν επιστρέψει στην Τουρκία, θα το ξαναπώ, μίλησα πριν για 468, οι περισσότεροι επιστρέφουν σε εθελοντική βάση. Και αρχίζει και ένα πρόγραμμα εθελοντικών επιστροφών προκειμένου να φύγουν από τα νησιά οι άνθρωποι αυτοί και να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους σε θελοντική βάση. Εννοείται ότι αυτό δεν θα ισχύσει για τους ίδιους οι οποίοι δεν πρόκειται να επιστρεφούν στη Συρία. Δουλεύουμε επίσης και συνεργαζόμαστε στενά με τις ελληνικές αρχές ώστε να μπορούν να υποδέχονται περισσότερους και σε καλύτερες συνθήκες. Ιδιαίτερα μας απασχολεί το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων και των πιο ευάλωτων ατόμων και προσπαθούμε με τις ελληνικές αρχές να τους βγάλουμε από τα hot spots τους ανθρώπους αυτούς. Έχει γίνει για τους ε, ασυνόδευτους ε, ανηλίκους. Κατά τα άλλα στην Άγκυρα έχουμε πρόσβαση, αντιπροσωπεία μας δηλαδή, στους καταβλισμούς όπου φιλοξενούνται οι πρόσφυγες και μπορούμε να επιθωρήσουμε την κατάσταση εκεί, να συζητήσουμε και να προτείνουμε και κάποιες διορθώσεις διαπιστώσαμε πολλές φορές ότι αυτοί οι οποίοι επιστρέφουν δεν γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους. Οπότε έχουμε ζητήσει από τις τουρκικές αρχές να ετοιμάσω κάποια εγχειρίδια, κάποια φυλάδια, στις γλώσσες των ανθρώπων αυτών με στοιχεία ώστε να ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους. Στην πρώτη τελευταία μου επίσκεψη συζήτησα με τον ε, υποδιευθυντή ενός κέντρου για τους μετανάστες εκεί και είδαμε πόσο σημαντικό είναι όταν επιστρέφουν στην Τουρκία από την Ελλάδα να βρίσκονται υποκαθεστώ προστασία. Για μα ήταν ζωτική σημασία σε αυτό. Οπότε, όπω είπα και από την αρχή, η συμφωνία κρατάει. Είναι εύθραυστη, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι λειτουργεί. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Τώρα, έχω εδώ έναν μακρύ κατάλογο ομιλητών. Θα σας διαβάσω τα ονόματα και μετά, αν κάποιος δεν περιλαμβάνεται... Mr. Coelho, Mr. Dupré, Mrs. Piri, as the rapporteur in AFET for Turkey, Mr. Niedermüller, Mrs. Pagazau Tundi Ruiz, Mr. Marianne, Mrs. Gomez, Mrs. Schlein, and Mrs. Keller. I read your name. Η κυρία Ινχετφέλτ επίση. Και εσεί, ναι. Καλώς. Η κυρία Σίπελ πρώτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να με ακρηγορήσω για να δώσω την ευκαιρία και στου υπόλοιπου να μιλήσουν. Καταρχήν, ε, θα ήθελα να πω ότι ένα πράγμα είναι εντελώ ξεκάθαρο. Ε, και έχουμε μια διαφορά από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια. Η Τουρκία ήταν έτοιμη να δώσει προστασία στους πρόσφυγες. Ε, αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά και είναι κάτι λυπηρό που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Δεν θα επανέλθω σε όλα τα ζητήματα που θέσατε, αλλά θα ήθελα να μου πείτε κάτι για τις συνεχιζόμενες εκθέσεις που λαμβάνουμε. Όχι μόνο ότι χτίζει ένα τείχος η Τουρκία, και όχι για να αποφύγει να έρθουν μέλη του ΆΙΣΙ στην Τουρκία, αλλά για να αποφύγει να έρθουν περαιτέρω πρόσφυγες στην Τουρκία. Και έχουμε επίση και εκθέσεις που συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ότι υπάρχουν πυροβολισμοί κατά των προσφύγων και οι πρόσφυγες πεθαίνουν, μάλιστα και παιδιά στα σύνορα. Μπορείτε να αναφερθείτε σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Κύριο Σκοέλιο. Όχι. Κύριος Δεπρέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Επιτροπή για την ενημέρωση. Δεν θα επανέλθω τώρα στις κρίσεις που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία. Απλώ να πω ότι σε σχέση με του στόχου που είχαν δηλωθεί από την Κομισιόν, τα αποτελέσματα τα έχουμε. Γιατί ο αριθμό των ελεύσεων έχει μειωθεί σημαντικά και ο αριθμό των νεκρών έχει μειωθεί σημαντικά επίση. Και αυτοί είναι δύο από του στόχου που είχαν τεθεί. Επίση, σημειώνω τα όσα είπατε. Δηλαδή ότι γενικώ σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, Υπάρχει εξέταση για το κάθε άτομο και υπάρχει και το θέμα της έφεσης. Απλώς θέλω να ρωτήσω αν αναστείλει τη διαδικασία η έφεση και θα ήθελα τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και έχω κάποιες ερωτήσεις τώρα. Είπατε ότι έχουμε 468 πρόσφυγες που στάλθηκαν πίσω στην Τουρκία από την Ελλάδα, αλλά είπατε ε, ότι ε, από την ίδια εποχή 546, δηλαδή πριν τη συμφωνία είχαν σταλεί περισσότεροι από τη μετά. Πίσω. Δεύτερον, σε ποια βάση επιστρέφονται, βάση της διμερούς συμφωνίας επαναπρόθεσης Ελλάδας-Τουρκίας ή βάση της συμφωνίας επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Θα ήθελα να μου πείτε ακριβώς πώς έχει η κατάσταση. Τρίτον, πάνω από τρία δις έχουν ε, προβλεφθεί από τη Συμφωνία και έχουμε 14 εκατομμύρια ευρώ για την ε, ακτοφυλακή ε, στην στο Αιγαίο. Επίσης προβλέπεται ένα κονδύλι 20 εκατομμυρίων επιπλέον. Αρκεί αυτό το κονδύλι. Υπάρχουν ε, και άλλα κράτη τα οποία έχουν την υποχρέωση να φιλούν τις ακτές και υποφελούνται από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως πρέπει να το χάρη η Ιταλία, η Ελλάδα. Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντεπρέ, κύριε Πύρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μορντή για την εισαγωγή σας. Εγώ συμφωνώ ότι έκανε πολλά η Τουρκία τουλάχιστον έκανε πολλά όταν τα κράτη-μέλη ζήτησαν από την Τουρκία να αναλάβει δράση. Τώρα, κάτι επικριτικό. Την προηγούμενη Κυριακή λάβαμε μια κοινοποίηση από το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τρεις γυναίκες, τέσσερα παιδιά και ένας άνδρας δολοφονήθηκαν. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τέτοιες καταγγελίες και η Human Rights Watch έκανε μια τέτοια καταγγελία πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά αυτά τα θέματα, δηλαδή υποθέτουμε ότι η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα και πρέπει να το διερευνήσουμε αυτό. Ε, το αρνείται ο Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία ότι έγινε κάτι τέτοιο, αλλά είναι αποδεικτεί αληθινό ποιε είναι οι συνέπειε για τη συμφωνία, για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Είδαμε και πάλι ότι συνελήφθησαν δημοσιογράφοι και περασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δυστυχώ κάτι τέτοιο συνεχίζεται στην Τουρκία ε, βάσει αυτού του αμφιλεγόμενου ε, τρομοκρατικού νόμου. Έτσι λοιπόν, ε, τι συμβαίνει τώρα σε ό,τι αφορά τις απαιτήσει για την απελευθέρωση θεωρήσεων. Τρίτο σημείο. Το σαφές μήνυμα στους μετανάστες είναι ότι το να μπείτε σε μία βάρκα και να ρισκάρετε τη ζωή σας στη διαδικασία δεν αξίζει ενώ μπορείτε να ακολουθήσετε τον ασφαλή οδό της μετεγκατάστασης. Τώρα, αν μιλάμε για 711 ανθρώπους, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ασφαλής οδός ε, αυτή τη στιγμή και η Κομισιόν ε, σκέφτεται να προωθήσει αυτή την πρόταση για τη μετεγκατάσταση. Την τελευταία ερώτηση για την Ελλάδα. Είδαμε ότι ε, η Επιτροπή Εφετών ε, απέρριψε ε, τις επιστροφές στην Τουρκία. Υπάρχει τώρα περίπτωση να αλλάξει η Ελλάδα αυτή την Επιτροπή Εφετών και με ποιο τρόπο. Επίσης υπήρχαν καταγγελίες ότι η μπλοκάρει την πρόσβαση των δικηγόρων στην ακροματική διαδικασία. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή, εκεί, αυτοί οι δικηγόροι που έχουν πελάτες στο Μόρια δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης πριν να περάσουν από την Επιτροπή Εφετών οι πρόσφυγες. Ευχαριστώ επόμενος ομιλητές. Κύριος Χόλτερ. ευχαριστώ. Τρία ερωτήματα. Μας ανησυχούν τα συμβάντα στα σύνορα της Συρίας και ακούμε όλο ένα και περισσότερο ότι σκοτώνονται άνθρωποι. Το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένο πόσα τέτοια συμβάντα έχουν υπάρξει και ποια είναι η επικοινωνία σας με την Τουρκία. Από την περιφέρεια Ρότσαβα ακούγεται ότι η προσωρινή κυβέρνηση θέλει την επιστροφή και εμπόδιο στέκεται σε αυτό η Τουρκία. Και τρίτο ερώτημα. Οι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, μάλλον αυτοί που πήγαν στην Ελλάδα, κατέφτασαν στην Ελλάδα πριν από τις 18 Μαρτίου, τι θα συμβεί με αυτούς, ποια είναι τα σχέδιά σας, πώς θα βοηθήσετε τους ανθρώπους αυτούς προκειμένου να ενταχθούν ενδεχομένως και αυτοί στο πρόγραμμα με την κατάσταση. Υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν για παράδειγμα να πάνε στην Πορτογαλία και δεν μπορούν παρά το γεγονός ότι η πορτογαλική κυβέρνηση έχει δηλώσει τη διάθεσή της να τους υποδεχθεί. Δεν μπορεί να γίνει κάτι ώστε να φύγουν κάποιοι άνθρωποι προς τα εκεί και άλλα κράτη-μέλη έχουν εκφράσει την προθυμία τους να υποδεχθούν και να φιλοξενήσουν πρόσφυγες, αλλά προφανώς ε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Μάζε. Η κυρία Αρούτς. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω για τα στοιχεία που μας δώσατε, αλλά για μας τα στοιχεία πρέπει να τα δούμε σε κάποιο πλαίσιο. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν κάποιοι από τους συναδέρφους σας μας λέγαν ότι οι διαδρομές εισόδου αυτών που φεύγουν από τον πόλεμο ή διώκονται, 80% είναι μέσω της ε, Λιβύης και της Αιγύπτου. Θα διπλασιαστεί, λένε, ο αριθμός των ανθρώπων που τελικά θα πνιγεί στη Μεσόγειο το 2016. Εσείς ναι, μας δώσατε κάποια αριθμητικά στοιχεία. Μας είπατε ότι μειώνονται οι είσοδοι στην Ελλάδα. Αλλά οι προβλέψεις λένε ότι οι διπλοί θα χάσουν τη ζωή τους το 2016 στη Μεσόγειο. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερον, μπορείτε να μας πείτε και κάτι για τους λόγους γιατί εφαρμόζεται, υλοποιείται η πολιτική αυτή συμφωνία με την Τουρκία τόσο καλά. Παρόλα αυτά ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία παραιτήθηκε. Και τι επιπτώσεις θα έχουν θα έχει τελικά η συνέχεια αν τα νούμερα αυτά και οι προβλέψεις αυτές για θανάτους στη Μεσόγειο επαληφθούν. Ευχαριστούμε κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, τα δικά μου στοιχεία είναι λίγο διαφορετικά και προκύπτουν από τα στοιχεία της ελληνικής κυβέρνησης. Με βάση τα στοιχεία του Μαΐου συγκρινόμενα με τον Ιούνιο, οι πρόσφυγες συνολικά στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 4.300 αυτό σημαίνει ότι γίνεται μία διέλευση η οποία είναι μεν αργή, αλλά επί της ουσίας ο αριθμός ο οποίος παραμένει στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεύτερον, δεν έχει γίνει τίποτε πρακτικά για όλους τους πρόσφυγες οι οποίοι έχουν έρθει πριν τις 18 Μαρτίου διότι οι μετεγκαταστάσεις που έπρεπε να έχουν γίνει είναι ελάχιστες τις ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα και ο κύριος Αβραμόπουλος και εδώ έχουμε την αντίφαση από τη μια η Πορτογαλία να ζητά να υπάρξουν περισσότερες μετεγκαταστάσεις και από την άλλη από την Ελλάδα να μην φεύγει κανείς. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Είναι θέμα γραφειοκρατίας, είναι θέμα ρυθμίσεων, αλλά επί του πρακτέου οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν και δημιουργούνται πλέον πάρα πολλές εντάσεις διότι είναι μεγάλος ο αριθμός των προσφύγων και παράνομων μεταναστών πλέον στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν μπορούν να φιλοξενηθούν. Υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στην Καβάλα, Φερρυπίν. Σημερινά δημοσιεύματα μπορώ να σας στείλω να τα δείτε τι γίνεται. Και πρέπει να υπάρξει επιτέλους εφαρμογή της διαδικασίας μετεγκατάστασης από την κυρίως Ελλάδα για αυτούς οι οποίοι έχουν έρθει πριν τη συμφωνία με την Τουρκία. Δεύτερον, σας ενημερώνω ότι σχεδόν όλοι πλέον κάνουν αίτηση ασύλου. Όλοι λένε ότι είναι πρόσφυγες. Είτε είναι είτε δεν είναι. Σημερινό δημοσίευμα και εκτίμηση που υπάρχει λέει ότι από τις 58.000 και κάτι που είναι συνολικά στην Ελλάδα πρόσφυγες και παράτυποι μετανάστες, οι 50.000 θα κάνουν αίτηση. Τρίτον, το Υπουργείο έβγαλε μία απόφαση 31 Πέμπτου και λέει ότι επειδή πάνε πολύ αργά οι διαδικασίες παροχής ασυλού, όσοι παίρνουν την προσωρινή κάρτα για την προστασία, από τέσσερες μήνες θα πλέον θα μένουν στην Ελλάδα έξι μήνες και αν δεν γίνεται σωστά η καταγραφή θα μένουν ένα χρόνο. Άρα πρακτικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην πράξη έχουν δικαίωμα παραμονή στην Ελλάδα για ένα έτος που σημαίνει ότι δεν λύνεται κανένα πρόβλημα στην εφαρμογή τώρα της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, διότι εγώ πηγαίνω συχνά σε όλα τα νησιά. Παρακολουθώ το θέμα. Στη Σάμο. Στη Σάμο λοιπόν υπάρχουν αυτή τη στιγμή 1.200 άτομα, εκ των οποίων οι 300 δεν έχουν κάνει καν αίτηση ασύλου. Γιατί παραμένουν αυτοί εκεί και δεν επαναπροωθούνται. Παραμένουν εκεί εδώ και αρκετούς μήνες. Ερώτημα πρακτικό. Δεύτερον, είχατε πει ως Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα στέλνατε τουλάχιστον 400 υπαλλήλους της υπηρεσίας ασύλου για να βοηθήσουν στη διεκπαιρέωση των αιτήσεων ασύλου. Τι έχει γίνει. Έχει φρακάρει το σύστημα, καμία αίτηση πρακτικά δεν προχωρεί και με τη διαδικασία αυτή που λέτε από τους 8.300 εγώ σας λέω ότι ούτε του χρόνου δεν θα έχει τελειώσει η διαδικασία. Διότι έχουν δικαίωματα οι άνθρωποι, κάνουν την αίτηση, έχουν δικαίωμα εφέσεως, αλλά από εκεί και πέρα με τόσους λίγους υπαλλήλου που υπάρχουν δεν πρόκειται να διεκπεριωθεί καμιά αίτηση. Άρα λοιπόν είναι επιτυχής η εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία γιατί κανένας δεν πάει πίσω. Και δεν πάει κανένας πίσω διότι δεν εξετάζονται οι αιτήσει τους. Και για μεν τους Σύρους η διαδικασία προχωρεί, για όλους τους άλλους που κάνουν αίτηση ασύλου θα μείνουν στην Ελλάδα εφόσον τους χορηγηθεί και όσοι είναι παράτυποι μετανάστες δεν επιστρέφονται καν. Άρα λοιπόν πρακτικά που βρισκόμαστε. Αν φύγεις είναι 10 seconds. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να τα δείτε τα πράγματα πολύ πρακτικά και να υπάρξει μία πίεση. Το κλειδί λέγεται μετεγκατάσταση από την Ελλάδα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να εφαρμοστεί τώρα. Πρακτικά να συμμετάσχετε κι εσείς, να πάρει η Πορτογαλία όσους θέλει από την Ελλάδα. Να δουν οι πρόσφυγες ότι εφαρμόζεται η μετεγκατάσταση. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Γκόμες. Κοιτάξτε, είναι γελίο να πούμε ότι η συμφωνία λειτουργεί. Όταν υπόθηκαν όλα αυτά, βλέπουμε ότι διπλασιάζονται οι ζωέ από χώρες όπως η Αίγυπτος, φυσικά, για να μην αναφέρουμε τι συμβαίνει μέσω της Αλβανίας. Και επίσης μπορεί στη Σμύρνη κάποια δίκτυα διοικητών να έχουν διελθεί, αλλά πήγαν αλλού φυσικά και μάλλον εκμεταλλεύονται περισσότερο του ανθρώπου και βγάζουν περισσότερα χρήματα. Τι λέει η Κομισιόν για την απόφαση των γιατρών χωρίς σύνορα να αρνηθούν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην είναι συνένοχοι σε αυτό το εξωφρενικό σχέδιο να παραδίδονται οι πρόσφυγες χωρίς να υπάρχει σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τη σύμβαση για του πρόσφυγες. Γιατί φυσικά βλέπουμε τι συμβαίνει με την Τουρκία αφενός. Η Τουρκία έκανε κάποια δουλειά για τους πρόσφυγες, ε, για μεγάλους αριθμούς, αλλά από την άλλη δεν υπάρχουν οι να θεωρήσουμε εμεί ότι είναι ασφαλής τρίτη χώρα η Τουρκία ποιες εθνικότητες μετεγκαταστάθηκαν από την Τουρκία, δηλαδή αυτοί 711 άνθρωποι, σε ποιες εθνικότητες ανήκουν. Και η Κομισιόν ε, τηρεί μητρό αυτών των ανθρώπων, ξέρει που βρίσκονται. Ή κάποια στιγμή θα μάθουμε ότι κάποιοι που ήθελαν να μετακατασταθούν εκούσια, δεν πήγαν εκούσια. Δηλαδή λέγεται ότι πήγαν εκούσια, αλλά δεν πήγαν εκούσια. Πίσω. Και κάποιοι και κάποιοι βρέθηκαν ε, παράνομα στην Ελλάδα και έχουμε και σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη μετεγκατάσταση. Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτή τη μετακατάσταση. Η δική μου χώρα, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, είναι μια χώρα που είναι έτοιμη να δεχτεί πρόσφυγες. Και το ξέρει και ο Τζο. Και εγώ εργαζόμασταν ε, για μια περίπτωση 400 γεζίτη. Τους ε, φέραμε σε επαφή, δεν ξέραμε που είναι, ήρθαμε σε επαφή με το άσωμα τις ελληνικές αρχές και για τρει μήνε δεν λειτουργεί τίποτα. Είναι εντελώ γελίο και οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να έρθουν στην Πορτογαλία και είναι έτοιμη η Πορτογαλία να του δεχτεί. Γιατί δεν λειτουργεί λοιπόν, δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Μία μέρα θα πάω εγώ εκεί ίδιο ε, να τους καταγράψω. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που μένουν σε αποθήκες. Γιατί εντάξει, ο καταβλισμός της ε, ε διαλύθηκε, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι τώρα μένουν σε σκηνές και σε αποθήκες και έχουμε καταγγελίες από τη ΜΚΟ που λένε ότι είναι παγιδευμένοι άνθρωποι εκεί, ότι ουσιαστικά εκεί που μένουν είναι σαν ε, ποντικοφολιέ, αρνούνται και ΜΚΟ να πάνε εκεί. Και για το θέμα των ανηλίκων. Εγώ όταν πήγα πριν δύο μήνες στην Ελλάδα μου είπαν οι αρχές ότι δεν είχαν ικανότητα να ασχοληθούν με τους μετανάστες. Τι κάναμε για να τους βοηθήσουμε να έχουν αυτές τις ικανότητες για τους ανηλίκους. Και τι γίνεται τώρα με τα hot spot, με την κράτηση στα hot spot. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ευχαριστώ. Κυρία Σλά. Ευχαριστώ. Μιλάμε για 8 ή για 11 πρόσφυγες που έχουν δολοφονηθεί στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Τουρκίας από τις τουρκικές αρχές ενώ προσπαθούσαν να περάσουν ε, τα σύνορα στην επαρχία του Ατάη. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Συρίας έχουμε 60 ανθρώπους που έχουν δολοφονηθεί από τις αρχές του έτους. Υπάρχουν ε, και αποδείξει. Δεν έχουν αρνηθεί αρχές την πυροβολή, αλλά λένε ότι έριξαν προειδοποιητικούς πυροβολισμούς. Θα θέλαμε ε, να λάβουμε απαντήσεις για το τι συμβαίνει και μας λένε ότι προσπαθούν να επαληθεύσουν τι συμβαίνει και θέλουμε να δούμε και ποιε είναι και οι συνέπειε αυτών των συμβάντων στην συμφωνία. Σύμφωνα με τον, με τον Guardian, είναι ουσιαστικά δύνατο φυσικά ποιο να εγκαταλείψει νόμιμα τη Συρία και πώ ε, θα ξεφύγουν από τον πόλεμο οι άνθρωποι αυτοί. Η Κομισιόν πιστεύει ότι η Τουρκία μπορεί πράγματι να θεωρηθεί ασφαλής χώρα υπό το φως αυτό του γεγονότα. Νομίζω ότι ένας και μόνο θάνατος αρκεί για να μην θεωρούμε τη χώρα αυτή ασφαλή για τους πρόσφυγες και ακούσαμε αυτή την εβδομάδα να αναφέρεται ως επιτυχής αυτή η συμφωνία. Ποιο είναι το μέτρο της επιτυχίας, ο θάνατος και τα δεινά να έρχονται, να πηγαίνουν κάπως πιο μακριά από τα δικά μας σύνορα εμείς ε, λέμε μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται. Αλλά βλέπουμε και τα παιδιά να προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και έχουν δικαίωμα οι άνθρωποι αυτοί σε δίθυν προστασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που είπαν ότι οι θάνατοι στα σύνορα της Συρίας πραγματικά πρέπει να επιφέρουν κάποιες επιπτώσεις και θέλω να μας πείτε τι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι αυτές. Πολλές ανησυχίες εκφράστηκαν σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στην Τουρκία. Θέλω να μάθω τι κάνει η Κομισιόν για να παρακολουθεί την κατάσταση εκείνων που έχουν επιστραφεί. Γιατί πιστεύω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Εσείς στέλνετε ανθρώπους πίσω. Και στη συνέχεια τι, τους, αφήσ τους αφήνουμε στη μοίρα τους. Τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Και ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι δεν είχαν τη, δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ασύλου, ούτε ε, να υπαχθούν σε καθεστώς ε, διεθνούς προστασίας. Είναι ελάχιστοι άνθρωποι που κατάφεραν να, το κάνουν αυτό. Οπότε η Κομισιόν τι σκοπεύει να κάνει προκειμένου να παρακολουθεί την κατάσταση εκείνων που έχουν επιστραφεί προκειμένου να μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι δεν έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους. Από την άλλη πλευρά, στο Αιγαίο, είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνουν σεβαστά τα ε, δικαιώματα ασύλου και να υπάρχει και μια διαδικασία έφεσης. Και αυτό δεν είναι σημαντικό μόνο για τη δική μας Επιτροπή, αλλά είναι σημαντικό και με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, είναι σημαντικό με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι ε, σημαντικό για όλες τις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά έχει ασκηθεί απαράδεκτη πίεση στην ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να αλλάξει τον τρόπο λειτουργία αυτών των ε, αρχών που δέχονται τις εφέσεις. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και έχουν καταλήξει στο ότι άνω του 90% των αιτήσεων τελικά είναι παραδεκτές γιατί πραγματικά αυτή η συμφωνία ε, με την Τουρκία δεν λειτουργεί ακριβώς επειδή η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα. Δεν μπορείτε να επιστρέφετε ανθρώπους σε αυτή τη χώρα γιατί οι επιτροπές αυτές έχουν κάνει τη δουλειά τους σωστά και παρόλα αυτά ασκείται πίεση στην Ελλάδα προκειμένου να αλλάξει σύνθεση των επιτροπών αυτών ώστε να ε, δημιουργηθεί μια σύνθεση των επιτροπών αυτών στην Ελλάδα που δεν θα, γίνεται, που δεν θα σέβεται τα ανθρώπινα και ατομικά δικαιώματα ε, των ανθρώπων αυτών. Θα δούμε αν στο μέλλον οι επιτροπές αυτές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τον νόμο, αλλά πρέπει να πω ότι η πίεση που ασκείται είναι απαράδεκτη. Και αυτό δεν έγινε μόνο από την Προεδρία και από τα κράτη-μέλη. Και η Κομισιόν είπε στις, ε, στην Ελλάδα, στις ανεξάρτητες αρχές που δρούν εκεί, ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα. Είναι απαράδεκτο αυτό. Μεταφέρετε σας παρακαλώ αυτό το μήνυμα. Είπαν οι συνάδελφοι και σχετικά με την πρόσφαση σε δικηγόρους στα hot spot. Ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Και είναι πραγματικά ανισχυτικό ε, να ακούμε ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ενδέχεται να εμποδίζει την πρόσβαση των ανθρώπων αυτών σε δικηγόρους. Και υπάρχουν και η ΕΑΣΟ και υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι ε, διαδικασίες ε, δεν είναι οι προβλεπόμενες. Πολλές αιτήσει μάλιστα απορρίπτονται από την ΕΑΣΟ με μια λογική copy-paste, χωρίς να γίνονται σεβαστά τα ατομικά δικαιώματα των ανθρώπων. Και έτσι οι, ε, οι ελληνικές αρχές καταλήγουν να μην μπορούν παρά μόνο να έρθουν και να επιβεβαιώσουν τις αποφάσεις που έχει πάρει ήδη η ΕΑΣΟ. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό και επειδή ε, πρόκειται να ανανεωθεί και η εντολή προς την ΕΑΣΟ θα πρέπει εμείς οι βουλευτές να εξετάσουμε με πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο τι ακριβώς ε, εντολή δίνουμε, σε ποιους ανθρώπους, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους και για τις ζωές τους και όχι απλά γενικά για τις μελλοντικέ προοπτικές τους, αλλά για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους. Και θα ήθελα να ακούσω μια απάντηση σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ η κυρία Ίνφαλτ. Δεν θέλει το λόγο. Ο κύριος Μπολιέζη. Ευχαριστώ. Έφτασα κάπως καθυστερημένα και δεν θα ήθελα να πω κάτι λανθασμένο. Βάσει των ε, δεδομένων ε, που ε, έχουν αναφερθεί. Από ό,τι φαίνεται η συμφωνία έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις εισρωές στην Ελλάδα, δηλαδή των ανθρώπων που φεύγουν από την Τουρκία, όμως δεν λειτουργεί σε ό,τι αφορά τις επιστροφές από την Ελλάδα. Νομίζω ότι αναφέρεται σε 460 ανθρώπους. Και θέλω να αναφερθώ και σε κάτι άλλο. Εσείς ε, είπατε ε, ότι έχουμε 711 μετακαταστάσεις από την Τουρκία στην Ευρώπη. Αν θυμάμαι καλά, προέβλεπε η συμφωνία την διατήρηση της σχέσης ένα προς ένα μεταξύ όσων ε, είχαν επιστραφεί από την Ελλάδα στην Τουρκία και από όσων μεταξύ των Σύρων ήθελαν να μετακατασταθούν στην Ευρώπη. Τώρα, τελευταία, μια τελευταία σκέψη αφορά ε, κάτι που είπε κάποιος συνάδελφος πριν από μένα, δηλαδή ότι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας έχει πραγματικά ωφέλη σε ό,τι αφορά ε, το μπλοκάρισμα της Βαλκανικής Οδούς, αλλά βλέπουμε αύξηση των διελεύσεων στη Μεσόγειο. Και αυτό ε, μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε αν έχετε κάποια σχετικά στοιχεία στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Τώρα τελειώσαμε με τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Τώρα θα δώσω το λόγο και πάλι στον προσκεκλημένο μας. Ακούσατε πολλά σχόλια, πολλές ερωτήσεις. Προσπαθήστε παρακαλώ να μας απαντήσετε σε όσο περισσότερες ερωτήσεις μπορείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την τουρκική πλευρά, πρέπει να σας πω ότι αν δεν μπορέσω να σας ικανοποιήσω όσον αφορά τις απαντήσεις μου, θα επανέλθω, αφού ρωτήσω τους συναδέλφους που είναι εκεί. Λοιπόν, θα αρχίσω με την κυρία Σίπελ όσον αφορά τους πυροβολισμούς που ακούσαμε ότι έγιναν σε βάρος κάποιων προσφύγων. Ήρθαμε σε επαφή με τις τουρκικές αρχές επ' αυτού, όπως είπατε κι εσείς, αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς αυτούς και δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τέτοιους ισχυρισμούς για πυροβολισμούς στα σύνορα. Εμείς με την αντιπροσωπεία μας στην Άγκυρα οργανώσαμε μια αποστολή στα σύνορα για να καταλάβουμε κι εμείς καλύτερα ποια είναι η κατάσταση εκεί. Με δύο λόγια αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σίγουρα δεν είναι η συστηματική πολιτική αυτή της τουρκικής κυβέρνησης. Δεν βρήκαμε κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι όντως αποθούνται οι πρόσφυγες. Η πρόσβαση όμως από τα σύνορα έχει περιοριστεί. Δεν είναι όπως ήταν στην αρχή της κρίσης. Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν λαθροδιακινητές που δρούν στην περιοχή και όντω υπάρχουν και επεισόδια. Είναι σαφέ ότι σε διάφορα συμβάντα έχουν υπάρξει πυροβολισμοί. Αλλά πρόκειται για τοπικά συμβάντα και δεν πρόκειται για μέρος μιας συστηματικής πολιτικής. Πάντως το θέσαμε και θα συνεχίσουμε να το θέτουμε και να παρακολουθούμε την κατάσταση εκεί από κοντά. Έρχομαι τώρα στο πώς επιστρέφονται στην Τουρκία οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό που ρώτησε ο κύριος Δεπρέ. Βάσει της συμφωνίας από την 4η Απριλίου μέχρι χτες το βράδυ ήταν 468. Επιστράφηκαν βάσει της διμερούς συμφωνίας επανεισδοχής Ελλάδας Τουρκίας. Υπάρχουν όμως και οι 5.000 οποίους αναφερθήκατε, αλλά ο πρώτος αριθμός, 468, είναι πόσοι επιστράφηκαν στην Τουρκία μετά τις 4 Απριλίου, ενώ οι 5.000 κλπ περιλαμβάνουν και αυτούς που από την υπηρετική Ελλάδα επιστράφηκαν στην Τουρκία από την αρχή της χρονιάς για τα 20 εκατομμύρια για την ε, Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. όντω είναι για να υπάρξει μεγαλύτερη ανακούφιση. Τους δίνουμε επιπλέον πλοία και δυνατότητε να σώζουν ζωές στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο γενικότερα. Αν υπάρχει περίπτωση που μια αντίστοιχη βοήθεια θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά και σε άλλα σημεία, θα το κάναμε και εκεί. Όσον αφορά τώρα την κατάργηση των θεωρήσεων, την ερώτηση της κυρίας Σπύρη, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν πέντε κριτήρια, συν δύο, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα αντικειμενικά, πιέζει ο χρόνος. Η Τουρκία τώρα πρέπει να δείξει ότι μπορεί να συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αυτά. Αν γίνει, βεβαίως θα ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Έρχομαι τώρα σε αυτό που ρωτήσατε για την ελευθερία έκφρασης. Μια στιγμή διακόπτη πρόεδρος. Παρακαλώ, ησυχάστε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουμε όταν υπάρχουν πηγαδάκια στην αίθουσα. Συνεχίζω. Γι' αυτό που είπατε για τη χθεσινή δίωξη δημοσιογράφων και σύλληψη. Είναι κάτι που η Κομισιόν παρακολουθεί από κοντά και είπατε εκπρόσωπος και αρμόδιοι για τα θέματα αυτά ενημερώθηκαν. Και πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε ότι η ελευθερία έκφρασης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μεγάλη σημασία στην ελευθερία αυτή έκφρασης. Αν δείτε την έκθεση που έχουμε ετοιμάσει για την κατάργηση των θεωρήσεων και την ε, συνέντευξη τύπου που δώσαμε, γίνεται ολοφάνερο ότι θέλουμε να αποφύγουμε καταστάσεις όπου ο ευρύς ορισμός για την τρομοκρατία οδηγεί στην σύλληψη και δίωξη ανθρώπων οι οποίοι χωρίς καμία βία εκφράζουν τις απόψεις τους. Στηρίζουμε λοιπόν τις οργανώσεις που έχουν τον ίδιο στόχο με μας. Κύριε Πύρη, θέσατε κι εσείς και άλλοι ζήτημα για το συνολικό αριθμό ατόμων που από τις 4 Απριλίου μετεγκαταστάθηκαν. 711 λοιπόν. Αυτό είναι ένα νούμερο το οποίο είναι παραπάνω από το σύνολο των μεταναστών που επεστράφηκαν 468 είναι βάση της συμφωνίας αυτής. Απλώς κάποια στιγμή σε θελοντική βάση έπρεπε να υπάρξουν επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε στις 7 Ιουνίου με τους Τούρκους ομολόγους μας για βάση των ε, κανόνων του παιχνιδιού και είναι ανάγκη να υπάρξει αξιολόγηση για να δούμε κατά πόσο αυτό το πρόγραμμα εθελοντικών επιστροφών μπορεί να ξεκινήσει ή όχι. Να δούμε ποιε είναι οι συνθήκε που επικρατούν δηλαδή, για να δούμε αν είναι εφικτό. Κύριε Γκόμε, εσεί θέσατε το θέμα τη εθνικότητα των 711 που μετεγκαταστάθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όλοι Σύριοι. Και επειδή πολύ αναφερθήκατε στην Πορτογαλία, πρέπει να σας πω ότι από τους 711, 11 έχουν ήδη μετεγκατασταθεί από την Τουρκία στην Πορτογαλία. Αναγνωρίζω ότι δεν ρωτήσατε ακριβώς αυτό, είπατε από την Ελλάδα, αλλά θα έρθω σε αυτό σε λίγο. Όσον αφορά τώρα την ερώτηση Βάιτενχοφ για το τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι βρέθηκαν στην Ελλάδα πριν από τις 18 Μαρτίου. Για όλους αυτούς τον οποίο ισχυρισμοί είναι αποδεκτοί, ότι δηλαδή πρέπει να χαίρουν προστασίας, τότε υπάρχει το πρόγραμμα μετεγκατάσταση, που δεν αποτελεί μέρο της συμφωνία της 18 η Μαρτίου, αλλά έτσι κι αλλιώς έγινε μεταφορά από τα νησιά στην υπηρετική Ελλάδα. Θέσατε και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για το τι γίνεται άπαξ και μία αίτηση θεωρηθεί αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές. Δεν σημαίνει ότι δίνεται και το άσυλο. Σημαίνει ότι πρέπει να ξαναδούμε την αίτηση αυτή σε επίπεδο ατόμου. Γι' αυτό και κρατάει πολύ διαδικασία. Για την ερώτηση της κυρίας Πάσας Δενούντα κατά πόσο αλλάζουν οι διαδρομές. Δεν έχουμε ενδείξεις προς το παρόν ότι από τη διαδρομή του Αιγαίου έχουμε περάσει στη Μεσόγειο. Στη Μεσόγειο η κατάσταση είναι η ίδια όπως και πέρυσι προς το παρόν. Δεν έχουμε δει καμιά μεγάλη μετατόπιση επίσης εθνικοτήτων. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι δεν είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο σε λεπτομέρειες. Απλώς λέω ότι προς το παρόν δεν βλέπουμε τέτοια μετατόπιση των ανθρώπων δηλαδή που διέσχιζαν το Αιγαίο τώρα να προσπαθούν να διασχίσουν την Μεσόγειο από αλλού πιο νότια. Με ρωτήσατε επίσης ποιες είναι οι συνέπειες της παρέτησης του πρέσβη μας στην Άγκυρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν συνέπειες και η αντιπροσωπεία θα συνεχίσει να παρακολουθεί καθημερινά την κατάσταση. Και είναι κάτι για το οποίο θέλω να σας δώσω λεπτομέρειες. Πράγματι, ελέγχουμε πολύ προσεκτικά και από κοντά το τι γίνεται με τους ανθρώπους που επιστρέφουν στην Τουρκία. Έχουμε πρόσβαση σε όλους τους καταβλισμούς, σε όλα τα κέντρα υποδοχής των ατόμων αυτών που επιστρέφουν από την Ελλάδα στην Τουρκία. Το προσωπικό, η αντιπροσωπεία μας παρακολουθεί την κατάσταση από κοντά. Είχαμε μάλιστα την ευκαιρία να διαπιστώσουμε από πρώτο χέρι και να μπούμε σε συζήτηση σε βάθος με τους Τούρκους συναδέρφους μας για αυτά που είδαμε και για αυτά που θα θέλαμε να διορθωθούν. Παράδειγμα, έλλειψη ε, πληροφοριών ενημέρωσης αυτών που επιστρέφουν και τα δικαιώματά τους. Δεν έχουν πάντα πρόσβαση σε διερμηνείς. Πολλές φορές οι διαδικασίες είναι περίπλοκες και αυτό το θέσαμε. Επίσης είπαμε ότι ακούμε ότι τους παίρνουν τα κινητά όταν φτάνουν. Αυτό έγινε γιατί υπήρχε νομοθεσία που λέει ότι τα ηλεκτρονικά ε, μηχανήματα από τα οποία μπορεί κανείς να βγάλει φωτογραφίες απαγορεύονται. Και η αλήθεια είναι ότι όλα τα τελευταίες γενιάς ε, τηλέφωνα έχουν τέτοιες δυνατότητες. Τα άλλα, με τα άλλα δεν υπήρχε πρόβλημα. Μπορούμε λοιπόν να πάμε όπου βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί και θα συνεχίσουμε την δυνατότητα αυτή να τη χρησιμοποιούμε και στη συνέχεια. Ρωτήσατε επίσης για τις εθνικότητες. Σας είπα ήταν όλοι οι Σύριοι, 711 δηλαδή, που ε, μεταγκαταστάθηκαν είναι όλοι οι Σύριοι. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση στους καταβλισμούς και τα hot spots στην Ελλάδα. Εμείς στηρίζουμε τις ελληνικές αρχές με δύο τρόπους. Πρώτον, δίνουμε οικονομική αρρωγή για να βελτιωθούν οι συνθήκες στους καταβλισμούς και δεύτερον, μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων, Έχουμε κινητοποίησει το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας για να στηρίξουμε την ε, ελληνική κυβέρνηση. Επίσης, όμως, βοηθούμε και με την ανάπτυξη των δικών μας ειδικών, της ΕΑΣΟ για παράδειγμα και άλλων, στους ίδιους τους καταβλισμούς για να βοηθήσουν επιτόπου. Για την ερώτηση όσον αφορά τους ανήλικους, και εσεί το θέσατε κυρία Γκόμες. Έχω ενημερωθεί ότι πηγαίνουν σε ειδικά κέντρα το οποία έχουν σχεδιαστεί για να είναι ακριβώς κατάλληλα για την φροντίδα των ανηλίκων για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ατόμων. Αν εσείς έχετε μια διαφορετική πληροφορία, σας παρακαλώ να μου δώσετε στοιχεία για να το κοιτάξουμε. Εργαζόμαστε και με το ECHR προκειμένου να ε, υπάρχει δυνατότητα και για περισσότερους. Τώρα γιατί δεν πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε, έτσι καλώς το βάρο στην Ελλάδα, στην επιρωτική Ελλάδα κυρίω, είναι τεράστιο. Και εμεί θα συνεχίσουμε να αποφελούμαστε από κάθε ευκαιρία που μας δίνεται να τους βοηθήσουμε. Έρχομαι στην κυρία Κέλλερ τώρα. Σα είπα ότι έχουμε πρόσβαση στα κέντρα, τα επισκεφτόμαστε, συζητάμε με τους ανθρώπους σε ατομική βάση. Θα λοιπόν ότι οι περισσότεροι οι οποίοι επέστρεψαν στην Τουρκία Κοιτάξτε, η εντύπωσή μας είναι γενικά θετική. Ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Θα σας δώσω παραδείγματα συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, ξέρω ότι από τους 31 Σύριους οι οποίοι επέστρεψαν στην Τουρκία από την Ελλάδα, οι 9 σε θελοντική βάση, και μου το επιβεβαίωσε και ο ΙΕΙ αυτό, δέχτηκαν να επιστρέψουν στη Συρία. Ξέρω ότι η μη Συρία από τους 411, οι 132 τώρα έχουν πάει, έχουν επιστρέψει στις χώρες καταγωγής τους. 132 από τους 411 έχουν επιστρέψει στις χώρες προέλευσής τους. Αν θέλετε μπορώ να σας δώσω την ανάλυση στην ε, γεωγραφική 40 Αυγανοί αλλά και 39 Πακιστανοί, 17 από το Μπαγκλαντές, 18 από το Ιράν. Μέχρι τώρα 25 από τους 411 έχουν ζητήσει διεθνή προστασία, 5 από το Κογκό, 5 από το Αφγανιστάν και τώρα είτε έχουν το δικαίωμα ή βρίσκ, ελεύθερες κυκλοφορίες ή βρίσκονται σε κέντρα. Γνωρίζουμε πού βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί και τους παρακολουθούμε σε ατομική βάση. Έρχομαι τώρα και στο θέμα της ασφαλούς τρίτης χώρας. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά πρέπει να σας πω ότι από τη δικιά μας την πλευρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επιστολή που έστειλε στις ελληνικές αρχές εκφράζει την ε, εκτίμησή της ότι η Τουρκία έχει καλύψει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ασφαλής τρίτη χώρα για επιστροφή ε, των προσφύγων από τις 4 Απριλίου μετά από την ε, ατομική εξέταση των αιτήσεων ασύλου στην Ελλάδα. Ότι τα άτομα αυτά μπορούν να επιστρέψουν στην Τουρκία που θεωρείται ασφαλής χώρα. Τώρα για την Επιτροπή Έφεσης. Στην έκθεσή μας που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα θα δείτε ότι λέμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή πηγόντως από την Ελλάδα προκειμένου αυτή να ενισχύσει τις δυνατότητές της επεξεργασίας των αιτήσεων ασύλου και εφέσεων σε ατομική βάση ώστε να τις επεξεργάζεται όσο γίνεται πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας κυρίως την έννοια της τρίτης ασφαλούς χώρας. Αυτό τονίζουμε. Επίσης ξέρουμε ότι οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να τροποποιήσουν την νομοθεσία τους παρετέρω, ώστε να έχουν μια νέα αρχή εφέσεων που να είναι υπεύθυνοι για τις δικαστικές αναθεωρήσεις των αποφάσεων. Εγκρίθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, από την Ελληνική Βουλή, 16 Ιουνίου η τροποποίηση αυτή του νόμου και σίγουρα θα παρακολουθήσατε τη συνέντευξη τύπου. Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος, ο ίδιος, καλωσόρισε την ε, ε, ενέργεια αυτή των ελληνικών αρχών επιταχύνουν τις διαδικασίες. Πάντως, Ποτέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ζήτησε από την Ελλάδα να τροποποιήσει την νομοθεσία της όσον αφορά τα σώματα εφέσεων. Πιστεύω ότι έτσι έχω καλύψει τις ερωτήσεις σας με εξαίρεση το σημείο εκείνο που έχει να κάνει με τον οργανισμό ΕΑΣΟ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει θέσει θέματα και ανησυχίες για την πρόσβαση σε δικηγόρους των ε, μεταναστών, των ατόμων αυτών. Αν έχετε στοιχεία να μου τα δώσετε παρακαλώ. Αυτά νομίζω ότι σας κάλυψα. Ευχαριστούμε κύριε Μορντή Ευχαριστούμε για τις λεπτομερείς απαντήσεις σας. Η γραμματεία μου ζήτησε αν μπορείτε να μας δώσετε τα αριθμητικά στοιχεία να τα μοιράσουμε, θα ήταν κάτι χρήσιμο. Τώρα θα περάσουμε στις ψηφοφορίες, γι' αυτό υπάρχει τέτοια κινητικότητα. Σας ευχαριστούμε εκ νέου και να περάσουμε στις ψηφοφορίες, συνάδελφοι. So, dear Συνάδελφοι, όπως είπα στην αρχή της συνεδρίασης, δεν θα ψηφίσουμε την έκθεση Χολμάιερ σήμερα. Αναβάλλεται για τις 27, πιθανότατα. Και θα περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία της ενίσχυσης των ελέγχων στα εξωτερικά σύμφωνα, σύνορα, σύμφωνα με τις ε, σχετικές βάσεις δεδομένων. Έκθεση Μακοβέη. Να ρωτήσω την εισηγήτρια αν θα ήθελε το λόγο. Όχι. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Έχουμε μία τροπολογία που έχει αποσυρθεί. Χθες το βράδυ αποσύρθηκε. Πρόκειται για την 77. Δεν θα ψηφίσουμε λοιπόν την τροπολογία 77. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Παράγραφος 1 τροπολογία 24 και τροπολογία 25. Πρέπει να ψηφιστούν μαζί. Έχουν να κάνουν με μια πλήρη απόρριψη. Άρχεται η ψηφοφορία. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Χρειάζεστε την κάρτα σας, μάλιστα. Διατηρώ ανοιχτή την ψηφοφορία και μπορείτε να προσθέσετε και τη δική σας ψήφο. Ωραία, λειτουργεί. Υπάρχει άλλο πρόβλημα. Το ECR έχει ένα υπεράριθμο. Κάποιος θα πρέπει να αποσύρει την κάρτα του. Παρακαλώ κυρία Σίμερ. Εγώ ξέχασα την κάρτα μου. Μπορώ να στείλω κάποιον να μου τη φέρει. Ναι, κάντε το παρακαλώ. Πέρασε τις προφορίες. Απορρίπτεται. Να περάσουμε στην τροπολογία 26, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 76, ονομαστική ψηφοφορία. Την έχει ζητήσει το ΕΛΚ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 78, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5, Άρχη η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 82. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 82. Ζητά μια διαγραφή. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Άρχεται ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 83. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 84. Άρχεται τη ψηφοφορία. Πέρας. Έχω και άλλη μία ψήφο. Να τη μετρήσουμε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 85. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 89. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 91. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. 13. Έναρξη. Λήξη εγκρίνεται. Τροπολογία 88, άρχεται ψηφοφορία. Συγγνώμη, καταπίπτει λόγω της 13. Πάμε στη συμβαστική 8, άρχεται ψηφοφορία, ονομαστική. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβιβαστική 6. Και πάλι ονομαστική και τμήματική ψηφοφορία για τη συμβαστική 6. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Τώρα το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε. Στην τροπολογία. Δεκαεπτά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 17. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 96. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 103. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 113. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 114. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Πάμε στην 117. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 100... Όχι. Τροπολογία 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 118. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 119 έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 120. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στα εκτιμώντα συμβιβαστική 1, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την ΑΦΕΤ 6. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Συγγνώμη. 49. Ψηφίζουμε για τη 49. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα, τροπολογία 47, έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Συγγνώμη, εγκρίνεται, διορθώνει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 3, έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική 4. Έχουμε εδώ ονομαστική ψηφοφορία για τη συμβαστική 4 και τμήματική ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Γκρίνεται και για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται τη ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται. Επομένως, πάμε στην τροπολογία 6, άρχεται την ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 57, άρχεται την ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 64. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 65. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 66. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 67. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Περνάμε στην ε, τροπολογία ΦΕΤ 8. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 69. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 70. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε Στροπολογία 72. Υπάρχει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 73. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 75. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε την απόφαση της έναρξης των διαπραγματεύσεων, ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Μακοβέη. Σας ευχαριστούμε για την προσελευσή σας, συνάδελφοι. So we will have to suspect. Θα πρέπει να διακόψουμε λοιπόν μέχρι τις 12 ε, παρατέταρτο. Γιατί χρειαζόμαστε να έρθει ο κ. Δε για το επόμενο σημείο. Θα συνεχίσουμε στις 12 παρατέταρτο.

Uh, uh, Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Τώρα θα ακούσουμε σχετικά με την κατάσταση στην, ε, στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις ε, διαδικασίες ποινικέ υποθέσεις για την νομική συνδρομή προς τους ανθρώπους που έχουν, που έχουν στερηθεί την νομική συνδρομή σε περίπτωση εντάλματος, ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντεγιόν και συνέχεια σε όσα άλλα μέλη της Επιτροπής θέλουν να ε, παρέμβουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή για την ε, οδηγία και τον σχετικό τριμερή διάλογο που διεξάγεται και χαίρομαι που έχουμε λίγο χρόνο για να ενημερώσω την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για τις εξελίξεις. Ξεκινήσαμε η Πολαντική Προεδρία με τα άρθρα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σε σύλληψης. Τα πράγματα εξελίχθηκαν σχετικά ομαλά στην αρχή της Προεδρίας και έτσι πήραμε θάρρος για να συζητήσουμε και τα άλλα θέματα της ε, οδηγίας που ήταν κάπως πιο επίμαχα και πιο δύσκολα. Νομική συνδρομή για υπόπτους και για κατηγορούμενους σε ε, ποινικές διαδικασίες γενικά. Όπως θα θυμάστε, ε, το Κοινοβούλιο κατέθεσε διάφορες ιδέες να ευθυγραμμιστεί η οδηγία αυτή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο ε, υπήρχαν ε, ζητήματα και για κάποιες πολιτικές ομάδες εδώ αλλά και για, τον, και για το Συμβούλιο. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει έντονα. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να βρούμε ε, μια μέση λύση που ε, με τη στέρηση της ελευθερίας πλάς. Ε, δηλαδή όταν έχει στερηθεί την ελευθερία σου θα πρέπει παρόλα αυτά να ε, λαμβάνεις νομική συνδρομή σύμφωνα και με την οδηγία για την πρόσβαση σε δικηγόρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι λέει το Συμβούλιο, τι συμβαίνει αν έχεις απλά μια, μια έρευνα σε κάποια ε, ήπια ας πούμε, υπόθεση ε, ακόμα βρισκόμαστε στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων αλλά νομίζω ότι μπορώ να πούμε να μπορώ να πω ότι θα βρεθούμε σε ένα καθεστώς ελευθερία στέρησης ελευθερίας ε, συν και πλην κάπου θα τα βρεθούμε δεν υπάρχει πλέον διαφωνία ε, όσον αφορά την συμπερίληψη κάποιων από τον κατευθυντήριων γραμμών ε, της Κομισιόν σχετικά με την ποιότητα της νομικής συνδρομής και για το πώς θα οριστεί ε, ένας έλεγχος στην περίπτωση της νομικής συνδρομής μπορεί κανείς να πει ότι αυτό δεν θα πρέπει να βρίσκεται μόνο σε σύσταση και πλέον υπάρχει συμφωνία επ' αυτού και το ζήτημα που απομένει είναι να βρεθεί η σωστή διατύπωση. Συνολικά ε, ε, εισερχόμαστε στην κρίσιμη φάση τις επόμενες μέρες. Σήμερα το απόγευμα θα ενημερώσω τους σκιώδεις για το τι συζητήσαμε σήμερα το πρωί με την Προεδρία. Τους παρουσιάσαμε τις ε, τελευταίες μας ανησυχίες σχετικά με, με το κείμενο και εκείνοι έχουν πλέον επιλέξει κάποια από τα ζητήματα που θα παρουσιάσουν ε, στην Κορεπέρ αύριο και θα συζητήσουν με τα κράτη-μέλη αν μπορούν να ακολουθήσουν τη δική μας, τις δικές μας προτάσεις την πορεία που χαράσουμε εμείς και ελπίζει η Προεδρία ότι θα τα καταφέρει συμπεριλαμβανομένων και κάποιων κρίσιμων σημείων που θα συζητηθούν σε βάθος σήμερα το απόγευμα με τους Χιώδης. Την Πέμπτη έχουμε τον τριμερή διάλογο και με τους σκιώδεις σήμερα το απόγευμα θα καθορίσουμε τη στάση μας στον τριμερή αυτόν διάλογο. Και ως εισηγητής εγώ θα πρότεινα να πάρουμε αυτό που ε, ήδη μας έχει προσφέρει το Συμβούλιο να τηρήσουμε δηλαδή να προσπαθήσουμε δηλαδή να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα επί αυτής της Προεδρίας να γίνει δηλαδή ο τελευταίος τριμερής διάλογος και στη συνέχεια να επανέλθουμε το συντομότερο δυνατό εδώ στην Επιτροπή για έγκριση. Για τα κράτη-μέλη θα γίνει, ε, θα γίνει κορεπέρ στις 30 Μαΐ, Ιουνίου για να οριστικοποιηθούν και οι εργασίες από τη δική τους πλευρά. Αν όλα εξελθούν έτσι, ελπίζω ότι η ψηφοφορία στην ε, ΛΥΜΠΕ θα γίνει ε, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ευχαριστώ κύριε Ντεγιόν. Ποιος θέλει το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Ωραία. Σας ευχόμαστε τότε καλή επιτυχία για τους συνεχιζόμενους τριμερείς διαλόγους. Και περνάμε στο τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη για σήμερα το πρωί, που είναι ανταλλαγή απόψεων Επιγραφή ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη 29η Ιανουαρίου 2016 του Ιγνάτσιο Κοράου για πιθανές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ξένων ανηλίκων στην Σικελία. Σύμφωνα με τον κανονισμό, αν δεν έχει υπάρξει απάντηση ή η απάντηση ήρθε με καθυστέρηση, το θέμα αυτό έρχεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Στις 17 Ιουνίου λοιπόν υπήρχε η προθεσμία, δεν ε, υπήρχε απάντηση μέχρι τότε, οπότε κύριε Κοράο έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, γνωρίζουμε όλοι, η Ιταλία και συγκεκριμένα η Σικελία υφίσταται εδώ και χρόνια πολύ ισχυρή μεταναστευτική πίεση. Είχαμε αξιοσημείωτη αύξηση της παρουσίας ασυνόδευτων ενηλίκων στο νησί. Σήμερα φιλοξενεί η Σικελία περίπου 4.500 ε, ανήλικους ελοδαπούς ε, και έχουν καθοριστεί δομικές ε, δομές και το κόστος κάθε μέρα για κάθε ενήλικο είναι περίπου 76 ευρώ, από τα οποία 45 ευρώ χορηγούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ τα υπόλοιπα πρέπει να πληρώνει τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει του απαραίτητου πόρου για να επιστηρίξει αυτό το κόστο και έτσι λοιπόν ε, δεν ε, μπορούν πλέον να φιλοξενηθούν οι ανήλικοι και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτές τις δομές δεν έχουν πληρωθεί εδώ και δέκα μήνες. Η λύση που προτείνει η Περιφερειακή Αρχή είναι να μειωθούν τα πρότυπα της φροντίδας έτσι ε, ώστε το κόστος ε, να καλύπτεται από τα 45 ευρώ που δίνει το κράτος. Ε, τώρα, η Κομισιόν γνωρίζει αυτή την κατάσταση και θεωρεί ότι είναι νόμιμη και παραδεκτή και επίσης πώς σκοπεύει να βοηθήσει την κατάσταση με πρόσθετους πόρους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κοράο. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Κομισιόν, κύριε Κόρας. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας αυτή. Όσον αφορά την καθυστέρηση της απάντησης, ζητούμε συγγνώμη. Υπήρξε ένα πρόβλημα για το ποιος αναλάμβανε την ερώτηση αυτή, εσωτερικά ζητήματα και γι' αυτό υπήρξε καθυστέρηση. Θα σας απαντήσω όμως τώρα. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε ενημερωθεί από τις τελικές αρχές για τις δυσκολίες αυτές στη Σικελία. Όμως, επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακα των συνθήκων, η Επιτροπή παρακολουθεί προκειμένου τα κράτη-μέλη να συμμορφώνονται προς τις υποχρώσεις τους όσον αφορά το κεκτημένο για το άσυλο και περιλαμβάνει το κεκτημένο αυτό θέματα προστασίας των ασυνόδευτων ανελίκων. Εάν είχαν υπάρξει ενδείξει για συστηματικές παραβιάσεις των υποχρεώσεων της Ιταλίας, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διευκρίνιζε το θέμα με τις Ιταλικές αρχές. Οι χώρες μέλη μπορούν να έχουν χρηματοδότηση από το ΑΜΙΦ, το Ταμείο για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη. Είναι εθνικά προγράμματα. Ε, οπότε η Ιταλία για την περίοδο 2014-2020 έχει το εθνικό της πρόγραμμα δηλαδή δράσεις για την ενίσχυση των συστημάτων υποδοχής η αναβάθμιση της στέγασης και ειδική αρρωγή για τους ασυνόδευτους ανήλικους. Επιπλέον υπάρχουν και προγράμματα τα οποία στηρίζουν τους ασυνόδευτους ανηλίκους με χρηματοδότηση από το ΆΜΙΦ. Υπάρχει για παράδειγμα τώρα ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόστηκε πέρσι και φέτος με 11,9 εκατομμύρια που έχει ως στόχο να βελτιώσει τις δυνατότητε ε, των Ιταλικών αρχών στην Ιταλία για την υποδοχή ασυνόδευτων ανηλίκων και κυρίως ε, εκεί όπου η ροή των μεταναστών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επιπλέον, οι χώρε μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλη οικονομική αρρωγή από τα Ευρωπαϊκά Διευθυντικά Ταμεία, το Επενδυτικό Ταμείο και ιδιαίτερα το Κοινωνικό Ταμείο και το Περιφερειακό, όπω επίση και εκείνο για τη βοήθεια στου πιο ευάλωτου. Επίσης το 2016 υπάρχει και πρόγραμμα εργασίας με προτεραιότητα για τα παιδιά και τη μετανάστευση, κυρίως για τους ασυνόδευτους ανηλίκους με χρηματο δότηση για την συνοδεία και κυδαιμονία των παιδιών αυτών, για ανάδοχες οικογένειες δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κοράου, έχετε να προσθέσετε κάτι, όχι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει στις 27 Ιουνίου, 3 με 6 και μισή το απόγευμα. Θα ψεφίσουμε κατά πάσα πιθανότητα εκείνο το απόγευμα. Ωραία, σας ευχαριστώ όλους και καλή σας όρεξη.